Ladies Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερησίας διάταξης μετά από αλλαγές που έγιναν στην αρχική ημερησία διάταξη, τα σημεία 10 και 12 διαγράφονται επειδή συζητήθηκαν στην έκτακτη συνάντηση Επιτροπή αυτή στο Στρασβούργο. Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος 20, το 13 θα πρέπει να συζητηθεί αμέσως μετά την ακρόαση, τώρα το απόγευμα, και το 4 θα πρέπει να ψηφιστεί μαζί με τις άλλες ψηφοφορίε αύριο στις 10 λαμβάνοντας υπόψη ε, τις ε, χρονικούς περιορισμούς που έχουν οι άλλοι συγητές. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, συνεπώς θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερισία διάταξη. Ανακοινώσεις. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι θα μας χρειαστούν κάρτες, οι κάρτες της ψηφοφορίας, θα ψηφίσουμε και σήμερα και αύριο. Τώρα που τα είπαμε όλα αυτά μπορούμε να περάσουμε στο σημείο υπαριθμών 3 που αφορά την ακρόαση για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2. Θα ήθελα να καλωσορίσω ανάμεσά μας τον κύριο Ρισάρ Κρόνο από το Παρίσι, τον κύριο Μπάτσιρε Τσεπέλακα από το Πανεπιστήμιο Γεκελόνιν, τον Μάρκ Σόκρο κύριο Στατίσκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε την Ευαγγουίνεφ, τον διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα αρπαγής παιδιών. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους μου να με συγχωρήσουν γιατί δεν θα μπορέσω να παραμείνω κατά τη διάρκεια όλης της ακρόασης. Η κυρία Τελεβό θα με αντικαταστήσει. Θα ήθελα τώρα να τη ζητήσω να αναλάβει την Προεδρία και να παρακαλέσω και τον κύριο Σακρόνα να πάρει το λόγο. Monsieur Krohn, on σας ακούμε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας και για την τιμή που μου κάνετε. Ευθήκατε να μιλήσω εγώ σήμερα για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α ή μπις, ανάλογα το λέμε. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν θα μιλήσω ως πανεπιστημιακός, αλλά θα σας ε, μιλήσω ως κάποιος ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής ε, σχολής ε, συμβολιογράφων στην Γαλλία και θα σας μιλήσω για την δικαιοδοσία από την ε, οπτική γωνία των συμβολεογράφων. Δηλαδή, ποιος είναι αρμόδιος για αυτή τη ε, δικαιοδοσία. αυτό, διότι αυτό είναι το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ε, συνήθως, διότι εμείς σχεδόν ποτέ δεν εμπλεκόμεθα σε θέματα που αφορούν γονική μέρημνα ή απαγωγή τέκνων εκτός της χώρας. Καταρχάς, το θέμα αυτό αφορούσε μόνο τα δικαστήρια και μετά πέρασε και στις δικαιοδοσίες των συμβολιογράφων. συμβολιογράφοι στις διάφορες διαδικασίες διαζυγίων στα διάφορα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στη Γαλλία επέτρεψε στους συμβολιογράφους να δουν με σαφήνεια και σε ένα πρώιμο στάδιο τι θα συνέβαινε με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού των Βρυξελών 2 όχι μόνο την ε, στιγμή του διαζυγίου, αλλά και τη στιγμή κατά την οποία πρέπει να παρέχει διάφορες συμβουλές ο συμβολιογράφος στους μελονύμφους, ε, ενδεχομένω ή σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να παντρευτούν κυρίως όταν είναι, έχουν δύο διαφορετικές εθνικότητες και προχωρώντας να φτάσουν ίσως και στις περιπτώσεις διαζυγίου μεταξύ δύο συζύγων. Έτσι λοιπόν, σε θέματα δικαιοδοσίας, βάσει αυτού του κανονισμού των Βρυξελών 2, βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες. Ρόλο συμβούλου λοιπόν, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Καταρχάς, σας είπα γιατί μπορέσει να συνταχθεί η σύμβαση γάμου και μετά σε περίπτωση διαζυγίου για να δοθεί η κατάλληλη συμβολή. Όταν γίνεται συμβουλή. Όταν ε, γίνεται το συμβόλαιο γάμου, ο συμβολεογράφος είναι αυτός ο οποίος θα δει με κάθε ε, έναν από τους μελονύμφους ποια είναι τα περιουσιακά του στοιχεία για να δει μετά κατά πόσον θα συνάψει ένα συμβόλαιο. Μετά, εάν θέλει κάποιος από τους δύο να έχει διευκρινήσεις για την ε, δικαιοδοσία, για το τι θα ακολουθήσει για το πώς ε, αν υπάρξει διαζύγιο θα μοιραστεί η περιουσία ε, είναι θέματα τα οποία μας αφορούν. Στην Γαλλία και όχι μόνο η επιλογή του νόμου που θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της ε, συνθήκης της Χάγης μπορεί κανείς να επιλέξει. Ξέρουμε ότι οι μελώνυφοι μπορούν από την θέσπιση και από την σύνταξη μάλλον του ε, συμβολέου γάμου να αποφασίσουν εάν θέλουν να τους εφαρμοστεί η νομοθεσία ε, του Παρισιού, της ε, Ολλανδίας, ακόμη και σε περίπτωση διαζυγίου για τα θέματα της διατροφής, ποια νομοθεσία θα εφαρμοστεί. Και βεβαίως μπορούμε να σκεφτούμε το ότι στο μέλλον η δικαιοδοσία και το καθεστώς που θα εφαρμόζεται θα μπορέσουν να δουν με πρακτικό τρόπο τη, την κατάσταση ώστε να μπορέσουν να διευκολυθούν οι διαδικασίες. Τώρα, στα πλαίσια της, του διαζυγίου, ο ρόλος συμβούλου του συμβολεογράφου είναι εξαιρετικά σημαντικός. Διότι από τη στιγμή κατά την οποία οι σύζυγοι αρχίζουν αυτή τη διαδικασία για να πάρουν διαζύγιο, πρέπει να εξηγήσουμε, να τους εξηγήσουμε ποιοι είναι αρμόδιοι για κάθε θέμα βάση του κανονισμού Βρυξέλλες 2 και να επιστήσουμε και την προσοχή τους στο ποιος είναι αρμόδιος, ποιος έχει την διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός Ρώμη 3 είναι ένας κανονισμός ο οποίος κάπως έχει αμβλύνει την διαδικασία, το θέμα τους ε, προσφυγής στην ε, ε, διαδικασία και την δικαιοδοσία είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε και με τρίτες χώρες. Και σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως στη Γαλλία, όταν το διαζύγιο αφορά ένα ζευγάρι γαλλοαγγλικό, στη, βουλεύουμε στην σύζυγο να ζητήσει να τις εφαρμοστεί το αγγλικό δίκαιο δεδομένου ότι δεν έχει ε, τέτοιου είδους ε, ε, ε, διατάξεις που να μην την δημιουργούν πρόβλημα. Είναι πιο απλά τα πράγματα και σε θέματα τη, κυρίως καταβολής διατροφής είναι πιο απλά και προς όφελός της. Τώρα, έτσι πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Υπάρχει μία μια δυσκολία όσον ε, αφορά το θέμα της εθελούσιας επιλογής δικαιοδοσίας. Υπάρχει αυτή η δυσκολία, ενώ είναι δυνατόν να επιλέξει κανείς όταν παντρεύεται ποιο δίκαιο θα ακολουθήσει, όταν παίρνει διαζύγιο πολλές φορές υπάρχει δυσκολία όσον αφορά την επιλογή της δικαιοδοσία. Κάποια κράτη δέχονται την ε, δυνατότητα να επιλέξει το δικαστήριο που έχει τη δικαιοδοσία ένας από δύο από τους συζύγους, ενώ σε άλλες ε, περιπτώσεις, ε, εάν μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα αντιπαλότητας δύο νομοθεσιών, αυτό είναι δύσκολο. Πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και τη δυσκολία αυτή. Να επιλέξουμε το δικαστήριο εκ των προτέρων και ευθύ εξ αρχή, ώστε σε περίπτωση διαζυγίου να μην υπάρχει πρόβλημα και να ξέρει ευθύ εξ αρχή ο κάθε σύζυγος τι θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση διαζυγίου. Εάν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να ε, βελτιωθεί εδώ η κατάσταση, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε στα πλαίσια του κανονισμού Βρυξέλλες 2 να γίνεται επιλογή του δικαστηρίου που θα έχει την δικαιολογία ή τη δικαιοδοσία, συγγνώμη, ή κατά τη διάρκεια της σύναψης του συμβολέου γάμου ή κατά τη διάρκεια του γάμου ή όταν υποβάλλεται η τη δικαιοσύνη ή κατά τη διάρκεια της σύναψης του συμβολαίου γάμου ή κατά τη διάρκεια του γάμου ή όταν υποβάλλεται συγγνωμη η κατα τη διαρκεια της συναψης του συμβολεου γαμου διαζυγίου. Και θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η εθνικότητα ή ο συνήθις τόπος διαμονής των συμβαλωμένων, των συζύγων θα μπορούσε να καθορίσει και την, ε, το αρμόδιο δικαστήριο σε εθελούσια βάση. Τα κριτήρια που ακολουθούνται είναι τα κριτήρια που ισχύουν στο κοινοτικό δίκαιο ώστε να μπορέσουν να επιληθούν οι διαφορές ε, ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα θέματα αρμοδιότητες, αρμοδιότητες είναι θέματα τα οποία υπάρχουν και σε άλλες νομοθετικές πράξεις ε, στην κοινωτική νομοθεσία. Γιατί δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να το προβλέψουμε και εδώ στα πλαίσια του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Δεν σας λέω τίποτα καινούριο, διότι τα κείμενα τα οποία μου υπευλήθησαν παρά το γεγονός ότι τα τελευταία έφτασαν μέσω του τηλεφώνου σήμερα το πρωί και ήμουν ήδη στο τρένο ε, μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο λέγω αποτελεί αντικείμενο πρότασης οι οποίες έγινε πολλές φορές και εγώ απλώς το επαναλαμβάνω. Τώρα, οι σύζυγοι θα πρέπει να προβλέπουν καλύτερα τις καταστάσεις. Ακόμη και για να διευκολυνθεί αυτός ο οποίος θα κληθεί να τους συμβουλεύσει όταν έχουν πρόβλημα. Τώρα, εάν μια τέτοια ρήτρα συμπεριληφθεί στην ε, την σύμβαση γάμου θα πρέπει να γίνει με πνεύμα ε, ε ειρηνικό θα έλεγα, διότι δεν σημαίνει ότι όταν κανείς παντρεύεται και κάνει συμβόλαιο γάμου πρέπει απαραίτητο να περάσει από τη δύσκολη φάση του διαζυγίου αργότερα. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό, εκ των προτέρων, και τα δύο μέρη θα μπορούσαν να καθορίσουν και να γνωρίζουν ποια είναι η αρμόδια δικαιοδοσία τη στιγμή την οποία θα θελήσουν, αν θελήσουν, να λάβουν διαζύγιο. Επίσης, σύμφωνα με την πρακτική, σας δίνω εδώ ένα παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε ότι και σε άλλες νομοθεσίε υπάρχει. στην Γαλλία οι συμβολιογράφοι πολλές φορές βρίσκονται σε δύσκολη θέση όταν πρέπει να συνάψουν συμβόλαια γάμου μεταξύ Γάλλου και Βρετανού πολίτη. Διότι η Βρετανία, από τη στιγμή που κάποιο έχει την εθνικότητα, μπορούν να επιλέξουν την νομοθεσία τους και ζητούν να έχουν ένα prenup, δηλαδή μία σύμβαση στην, ε, που, να έχει ισχύ στη Μεγάλη Βρετανία και περίπου ε, την ίδια σύμβαση στην ε, Γαλλία. Έχουν λοιπόν αυτή την επιλογή μεταξύ των δύο. Οι Βρετανοί λοιπόν επιβάλλουν μία ρήτρα επιλογής δικαστηρίου και δικαιοδοσίας αρμόδιας τη στιγμή που κάνουν αυτό το προγαμιαίο συμβόλαιο. Και πολλές φορές σε άλλες περιπτώσεις ε, η ρήτρα αυτή ε, είναι μια ρήτρα την οποία δεν συμφωνούν πάντα να συμπεριλάβουν στα διάφορα προγραμμία συμβόλαια οι συμβολεογράφοι, διότι είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στα πλαίσια του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Η νομολογία η γαλλική όσον αφορά την ευθύνη του συμβολεογράφου ορίζει ότι ο ρόλος του συμβολεογράφου είναι συμβουλευτικός και δεν μπορούν στα προγαμιαία συμβόλαια να συμπεριλαμβάνονται ρήτρε οι οποίες δεν προβλέπονται στην γαλλική νομοθεσία. Γι' αυτό πολλές φορές πρέπει να πω ότι αρνούμεθα να παρέμβουμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και να συμπεριλάμε στα προγαμιαία συμβόλαια τέτοιου είδους ρήτρες. Θα ήταν λοιπόν πραγματική πρόοδος, καινοτομία, εάν ε, η εξουσιοδότηση να επιλέγει καλής ε, την ε, διεθνή δικαιοδοσία, το αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή σε περίπτωση του θα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί εδώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, πολύ. Για την Κάνατε αναφορές και στην καθημερινή ζωή να περάσουμε στον επόμενο μιλητή, που είναι ο κύριος ε, Τσέπελάκα. Ειλικρινά με ευγνώμων που με προσκαλέσατε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου ζητείτε και να μιλήσω για θέματα εφαρμογής ε, μετά από τη λήψη αποφάσεων για την γονική μέρευνα. Δίχω άλλο δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναφερθώ σε αυτά τα πολύπλοκα θέματα σε 20 λεπτά. Εκτός από αυτό έχω πόλη τη συνέστηση ότι τα πολλά, τα πολυάριθμα προπαρασκευαστικά έγγραφα που σας έχουν δοθεί φύγουν λεπτομερώς το πρόβλημα. Οι απαντήσεις που οι χώρες μέλη στέλνουν απαντώντας τα ερωτηματολόγιο που ε, συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέρουν να δώσουν μια γενική εικόνα που αφορά τη μη αναγνώριση και τη μη εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τη γονική ευθύνη. Για τους λόγους αυτούς, αυτούς και για να μπορέσω να συμβάλλω στο έργο σας, δεν θα επαναλάβω τα όσα έχουν ήδη υποθεί και λεχθεί αλλού. Αντίθετα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα προβλήματα που κατά την άποψή μου είναι κεφαλαιόντου σημασίας για την αξιολόγηση του προγράμματος εφαρμογής σύμφωνα με τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσω την περίπτωση Boys κατά Δίες, η οποία πρόσφατα, για την οποία πρόσφατα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η περίπτωση αυτή αποφασίστηκε, για την περίπτωση αυτή λήφθη απόφαση την 9η Σεπτεμβρίου 2015 και αφορούσε την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις αποφάσεις που αφορούσαν τη γονική ευθύνη. Θα αναφερθώ σε μερικά προβλήματα με βάση ε, την ανάλυση που έκαναν τα αρμόδια δικαστήρια με βάση τα άρθρα 28-29 του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Το πρόβλημα της εφαρμογής αυτών των ε, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ε, Μιλάμε λοιπόν ε, για αυτές ε, τις ε, καταβολές και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλά εθνικά συστήματα παρέχουν διάφορα μέτρα που έχουν σκοπό στοχεύουν στη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο κύριος Βόες και η κυρία Βέτς παντρεύτηκαν στο Βέλγιο το 1997 και απέκτησαν δύο παιδιά. Διαζεύτηκαν το 2005 και η κυρία Βίες πήγε στη Φιλανδία. Το 2007 το δικαστήριο στη Γάνδη έλαβε απόφαση σε ό,τι αφορά την επιμέλεια, την κατοικία, το δικαίωμα πρόσβασης <coughs> και την συντήρηση των παιδιών. Το δικαστήριο συμπλήρωσε την απόφασή του με επιβάλλοντας και μια χρηματική ποινή έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τα δικαιώματα πρόσβασης που θα είχε ο κύριος Μπόες. Το ποσό αυτό ήταν 1000 ευρώ παιδί. Ορίστηκε στα 1000 ευρώ αναπαιδί. που θα έπρεπε να πληρώνεται στον κύριο Μπόεση για κάθε μέρα που την παιδί θα ήταν παρόν. Το ανώτατο ποσό του ποσού αυτού ορίστηκε στις 25.000. Ο κύριος Μπόες απευθύνθηκε στα φιλανδικά δικαστήρια και ζήτησε να ληφθεί μια απόφαση που τα απαιτούσε από την κυρία Βίεζα να του πληρώνει αυτό το ποσό που αποφασίστηκε από το Βελικό Δικαστήριο το 2007. Από άποψη νομική θέτει ορισμένα θέματα. Όσοι σα ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Στην περίπτωση που ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με τρία προβλήματα. Καταρχάς, Υπήρχε αμφιβολία σχετικά με το κατά πόσον θα έπρεπε το αίτημα του κατηγορού να, κατηγορηθεί, να θεωρηθεί ε, ως ένα οικονομικό αίτημα. αν συνέβαινε το πρώτο θα σήμαινε ότι αυτό δεν εμπίπτει ε, στον, στα, στα πλαίσια του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Αυτό όμως ήταν αναγκαίο μόνον για να μπορέσουν να εφαρμοστούν δύο μέτρα εφαρμογής και συγκεκριμένη αυτή η περίπτωση ήταν σχετικά απλό. Το δικαστήριο, δικαστήριο ακολούθησε την άποψη του δικαστή Σκούναρ και αρνήθηκε να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα αναφέροντας ότι οι χρηματικές ποινές είναι συμπληρωματικές στη βασική υποχρέωση, στη βασική διατροφή. Γιατί εδώ στόχος είναι να διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα πρόσβασης που είχε δοθεί στην ίδια απόφαση θα είναι αποτελεσματικό. Αυτό ασκεί οικονομικές πιέσεις στο πρόσωπο εκείνο που έχει αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού έτσι ώστε να συνεργάζεστε προκειμένου ο πατέρας να μπορεί να βλέπει τα παιδιά του, να έχει δικαίωμα πρόσβασης. Το δικαστήριο κατέληξε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το ποσό αυτό είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο το οποίο χρησιμεύει για να προστατεύσει ένα δικαίωμα το οποίο δεν εντάσσεται στα πλαίσια του κανονισμού 44-2001 και όχι στα πλαίσια του κανονισμού 21-2201. Δεν εντάσσεται στο πρώτο κανονισμό, εντάσσεται στο δεύτερο. Το δεύτερο πρόβλημα δεν ήταν τόσο απλό, γιατί αφορούσε περισσότερο προηγμένα επίπεδα εξειδίκευση. Αν μία ποινή, μία, ε, ε, ένα τίμημα χρηματικό που καταβάλλεται αποτελεί μόνο το συμπληρωματικό μέτρο που αποσκοπεί στην εφαρμογή μιας απόφασης, τότε το ερώτημα είναι τι θεωρούμε γονική μέρημνα και, τι θεωρούμε, ε, και πώς θεωρούμε ότι εφαρμόζεται. Εδώ μιλάμε για ένα ποσό που επιβάλλεται και είναι αποτέλεσμα μια δικαστική απόφαση. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι βέβαιο κατά πόσο το περιεχόμενο αυτή τη ε, απόφαση θα πρέπει να έχει το ίδιο νομικό καθεστώ. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα επιμέλειας, την κατοικία του παιδιού και το δικαιώματα ε, πρόσβασης στο παιδί, όλα αυτά είναι θέματα γονικής μέρημνας. Και ως τέτοια θα πρέπει να αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται. Αντιθέτως, Μία ποινή, χρηματική ποινή, είπαμε ότι είναι συμπληρωματικό μέτρο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί διαδικαστικό θέμα, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο του δικαστηρίου, εκεί που θα πρέπει να γίνει και εφαρμογή. Υπάρχουν και ορισμένα βασικά θέματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για αυτό το συλλογισμό. Τα δικαιώματα που προκύπτουν από την γορική μέρημνα είναι η ουσία τα μέτρα που υιοθετούνται να διαφυλάξουν αυτά τα δικαιώματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ένα θέμα διαδικαστικό. Τα μέτρα αυτά εξαρτώνται από την απονομή της δικαιοσύνης ε, και από τους φορείς που την απονέμουν δικαστήρια, ε, αξιωματική δίωξη, ε, δικαστικοί κλητήρες κτλ. Το θέμα είναι κατά πόσο το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της χώρας όπου θα εφαρμοστεί η απόφαση θα μπορεί να εφαρμόσει το μέτρο αυτό που περιέχεται στην απόφαση που ελήφθη στην άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα διεθνούς οικογενειακού δικαίου. Αφορά το, το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του. Είναι ένα θέμα με το οποίο, το οποίο έχει απασχολήσει και άλλες νομοθεσίες. Ας ρίξουμε μια ματιά στο Διεθνές Δίκαιο των Υποχρεώσεων. Προκύπτει από το άρθρο 18.2 του κανονισμού Ρώμη 1 ότι η εγκυρότητα μιας σύμβασης μπορεί να αποδειχθεί από οποιοδήποτε τρόπο, είτε lex contractus είτε lex loci actus, υπό τον όρο ότι αυτός ο τρόπος απόδειξης θα μπορούσε να δοθεί από το δικαστήριο. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι ιδιαίτερα σημαντικό το κατά πόσον θα μπορούσε να ληφθεί μια απόφαση δικαιωτική μέρημνα από το νομικό σύστημα μιας χώρας όπου θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση. Παρόλα αυτά η ουσία του προβλήματος δεν βρίσκεται στα δικαστήρια, αλλά σε άλλους φορείς που είναι σημαντικοί για την καθημερινή ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν αρκετό να αναφερθούμε σε δύο θέματα, στη γλώσσα και την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με διασυνοριακή γονική μέρημνα, είναι σημαντικό, ανεξάρτητα από το παιδί, μπορεί να μάθει, ε, να γνωρίζει τις γλώσσες, είναι σημαντικό για το παιδί ε, να γνωρίζει τη γλώσσα και των δύο γονιών για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχει επαφή μεταξύ του γονιού και του παιδιού. Θα ήθελα να παραθέσω ένα πρακτικό παράδειγμα ενός Ιταλού πατέρα που έρχεται δύο φορές το μήνα στην Πολωνία για να επισκεφτεί την κόρη του που ζει με την Πολωνίδα μητέρα της. Ο πατέρας προσπαθεί να μάθει πολωνικά, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, ενώ η μητέρα δεν επιτρέπει στην κόρη της να μάθει ιταλικά. Η απόφαση του δικαστηρίου είπε ότι ο πατέρας θα συναντάται με την κόρη του ενώπιον ενός επιμελητή, κουράτορ. Το δικαστήριο όμως δεν είπε αν θα έπρεπε να παρίσταται και να σε μεταφοραστής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ολισμένες χώρες όπου οι διοικητικές αρχές απαγορεύουν την επικοινωνία με τα παιδιά στη μητρική τους γλώσσα εάν δεν είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά την παροχή ιατρικής φροντίδας, ένα θέμα που στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, εντάσσεται στα πλαίσια των ευθυνών και των δύο γονιών του 12χρονου κοριτσιού. Η μητέρα ήθελε να κάνει εξαγωγή εξαγωγή στα υγιή δόντια της κόλλης και για λόγους αισθητικούς να εμφυτεύσει άλλα δόντια. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι το να προβάλλει κανείς αντιρρήσεις σε μια τέτοια θεραπεία. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις που έχουν σχέση με γεγονότα που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης έχουν σημαντικές νομικές επιπτώσεις γιατί όπως προκύπτει από το άρθρο 47.1 του κανονισμού Βρυξέλλες 2α, η διαδικασία εφαρμογής διέπεται από το νόμο της χώρας ε, κράτους εφαρμογής. Το... Στην ουσία όμως, ε, ε, αν υπάρχει το θέμα της καταβολής του ποσού, θα σημαίνει ότι του ανούμετα να μπορέσουν να παραστούν σαν ε, και να πάρουν μέρο σε αυτές τις αποφάσεις. Τώρα, να πάρουμε στην περίπτωση που είναι σημαντικό να πούμε ότι και το βελγικό και το φιλανδικό δίκαιο επιτρέπουν στα δικαστήρια να επιβάλλουν ε, την καταβολή αυτού του ποσού. Η άμεση επίπτωση της ε, διαδικαστικής καταβολής ε, του ποσού αυτού το καθιστά μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Το δικαστήριο δεν έφτασε μέχρι σε αυτό το σημείο, αλλά ανέφερε το κίνδυνο του να γίνει μια διάκριση μεταξύ του δικαιώματος πρόσβασης ως έχει και της καταβολής του ποσού που το εξασφαλίζει. Αυτό προκύπτει από την απόφαση όχι ε, ένα ποσό το οποίο ε, αποφασίζεται από το δικαστήριο ενός κράτου μέλους αποτελεί μέρος του ίδιου πλαισίου εφαρμογής μιλώντας πάντοτε για τα δικαιώματα πρόσβασης και συνεπώς θα πρέπει να θεωρηθεί εφαρμοστέο σύμφωνα με τους κανόνες του Βρυξέλλες 2α. Με άλλα λόγια, η καταβολή του ποσού αυτού δεν θεωρείται θέμα διδικαστικό, αλλά θέμα ουσιώδες και αποτελεί μέρος του δικαιώματος επικοινωνίας ή πρόσβασης. Παρόλα αυτά, επιλύοντας το δεύτερο πρόβλημα, το δικαστήριο, κατέληξε στο τρίτο σημείο που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του βελγικού και του φιλανδικού νόμου. Σύμφωνα με αυτόν, ο δικαιούχος αυτής της πληρωμής δεν χρειάζεται να στραφεί προς το δικαστήριο για έναν τελεσίδικο ορισμό του ποσού ε, της καταβολής. Σύμφωνα με το φιλανδικό δίκαιο που πιστεύω και πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες μέλη, ο δικαιούχος θα πρέπει να ζητήσει από το δικαστήριο να ορίσει το τελικό ποσό της ε, ποινής, ε, της χρηματικής ποινής. Το πρόβλημα αυτής της διαφοράς επιλύθηκε δια της ε, αναλογίας με αναφορά στον κανόνα του άρθρου 49 της ε, κανονισμού Βρυξέλλες 1 ότι ένας πρώην, μια πρώην απόφαση, μια, μια ξένη απόφαση η οποία ζητά μια περιοδική καταβολή η οποία θα έχει τη μορφή ε, τιμωρίας θα πρέπει να εφαρμοστεί στη χώρα μέλος στην οποία γίνεται η εφαρμογή μόνον εάν το ποσό έχει τελεσίδικα αποφασιστεί από τα δικαστήρια της χώρας μέλους προέλευσης. Παρόλα αυτά, στην ε, απόφαση εδώ αναφέρθηκε ότι μόνο το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για θέματα επικοινωνίας μπορεί να ορίσει το ποσό του σχηματικής ποινής. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει διαδικαστικά μέσα έτσι ώστε να, να καταλήξει σε ένα τελικό ποσό, να πετύσει είναι να οριστεί το τελικό ποσό. Ακόμα λοιπόν και αν σύμφωνα με το νόμο του κράτους προέλευσης ο τελικός ορισμός της, ε, του ποσού αυτού δεν είναι αναγκαίος, θα πρέπει να εφαρμοστεί κάπου αλλού. Και γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να, συζητήσουμε την περίπτωση αυτή εδώ. Πιστεύω ότι η λογική του δικαστηρίου δεν αφορά μόνο την καταβολή αυτού χρηματικού ποσού. Θέλει να έχει μια ευρύτερη προοπτική σε ό,τι αφορά την, ε, τον οικογενειακό βίο. Είναι σαφές ότι αυτό βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Σαφώς προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου ότι οτιδήποτε αφορά τη γονική μέρημνα θα πρέπει να απασχολεί το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία και όχι το δικαστήριο εφαρμογής. Παρόλα αυτά το δικαστήριο ήταν γνώση των διαφορών μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών και επέμενε για τον αναγκαίο μηχανισμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυπταν. Αυτό που είναι σημαντικό προκύπτει από την απόφαση του Κατσιστηρίου ότι από τη στιγμή που η αρμοδιότητα για την ουσία της περίπτωσης μετατίθεται σχεδόν καθ' ολοκληρία στο δικαστήριο προέλευσης, το νομικό σύστημα της χώρα προέλευση θα πρέπει να λάβει αυτή την απόφαση, κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια άλλη χώρα μέλο. Κατά κάποιο τρόπο δείχνει την αλλαγή του παραδείγματος. Μέχρι τώρα μόνον μερικοί ε, ε, μίλησαν για θέματα ε, διαιτησίας. Παρ' όλα αυτά η διαιτησία ε, είναι καθήκον του δικαστηρίου προέλευσης να λάβει ε, υπόψη αυτό ότι η απόφαση του δηλαδή θα είναι δεσμευτική όχι μόνο στην, σε αυτή τη χώρα αλλά και σε άλλες χώρες μέλη. Κατά τον ίδιο τρόπο όσο πιο πολύ εμπιστοσύνη δίνεται στα δικαστήρια από μια χώρα μέλος τόσο πιο ε, υπεύθυνα καθίστανται σε ό,τι αφορά τα νομικά συστήματα άλλων χωρών μελών. Και επιτρέψτε μου να τελειώσω την παρουσίασή μου με δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς υπάρχουν πολλοί τρόποι για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις σε μία χώρα μέλος. Κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε μία ειδική διαδικασία. Μπορούσε να γίνεται με ή άνευ εξεκουάτουρ εκτελεστέο. Ε, θα μπορούμε να φανταστούμε τι συνέβαινε όπως κάνουν πάρα πολλοί μελετητές. Θα μπορούσαμε παρόλα αυτά να χρησιμοποιήσουμε πολλές λύσεις, αλλά ό,τι και να κάνουμε, όποια και είναι η επιλογή μας, η απόφαση θα πρέπει τεχνικά να είναι εφαρμόσιμη. Δηλαδή θα, μπορεί, θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζεται από τις αρχές διαφόρων νομικών συστημάτων. Και δεύτερον, το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στα δικαστήρια. Είναι πρόκειται για δασκάλους, ε, για διευθυντές ε, νηπιαγωγείων ή σχολείων, για γιατρούς ε, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις αποφάσεις ενός δικαστηρίου. Ανεξάρτητα από το μηχανισμό εφαρμογής που έχετε σκοπό να επιλέξετε, έχετε στο νου σας και αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Τσεπελάκ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνεισφορά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόν, ο οποίος ήρθε από το Παρίσι στις Βρυξέλλες για να μας κάνει την παρουσίασή του και από ό,τι κατάλαβα πρέπει να φύγετε στις 4. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιστροφή στο Παρίσι. Μπορώ να σας υποβάλω μια ερώτηση πριν φύγετε, παρακαλώ. Είπατε ότι είναι καλύτερα για την σύζυγο να αποφασίσει όταν κάνει το προγαμιαίο συμβόλαιο αν θα ακολουθήσει το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Όχι, όχι, όχι. Ε, δεν υπάρχει το ε, προγαμιαίο συμβόλαιο για τον ε, χωρίσει την ε, περιουσία ο κάθε σύζυγος όπως κάνουμε στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και μπορεί ο δικαστής στη Μεγάλη Βρετανία να αποφασίζει πώς θα γίνει η μοιρασιά των περιουσιακών στοιχείων. Τώρα, δίδονται διάφορες ε, αποζημιώσεις, αντισταθμίσματα στην σύζυγο που χωρίζει. Τα πράγματα σε εμά είναι διαφορετικά. Υπάρχει το καθεστώς που διέπει όπως και στο Βέλιο και στη Γερμανία και στην Ιταλία το προγραμμιό συμβόλαιο και το συμβόλαιο που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο αυτό και ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να το σεβαστεί. Και μετά ε, ο δικαστής μπορεί να κάνει διάφορες αναπροσαρμογές ώστε να μην ε, βλάπτεται υπερβολικά ο ένας από τον, σε σχέση με τον άλλο. Και βεβαίως αν ξανακάνει τη ζωή της η σύζυγος υπάρχει και ε, μνήα για το τι ακριβώς προβλέπεται για τα παιδιά. Πολλές φορές λοιπόν βλέπουμε η σύζυγος ενός γνωστού τραγουδιστή η επιχειρηματία να παίρνει 20 εκατομμύρια ευρώ μετά από 6 μήνες γάμου για όλα τα δικαιώματα δικαστής. Το είπα αυτό για να πω ότι υπάρχει μία ανισότητα και εγώ ως συμβολιογράφος Γάλλος όταν έχουμε να κάνουμε με Βρετανή σύζυγο της λέω αμέσως πηγαίνετε να δείτε ποια είναι τα δικαιοδοτικά δικαστήρια στη Μεγάλη Βρετανία για να έχετε καλύτερη αποζημίωση εάν ε, πάρετε διαζύγιο από ό,τι θα σας δώσει το γαλλικό δίκαιο. Και βεβαίως αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί από τη στιγμή που το λέμε αυτό στη σύζυγο, τη λέμε πηγαίνετε γρήγορα, διότι αν ε, ο σύζυγός σας προσφύγει πρώτα απ' όλα στη γαλλική διαδικασία, σύμφωνα με το Βρυξέλλες 2, θα προλάβει να σας επιβάλλει το γαλλικό δίκαιο. Πολλές φορές ε, πολλά άτομα αγνοούν τι απορρέει από την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Και ακόμη και αυτοί οι οποίοι το ξέρουν συμβουλεύουν τους πελάτες τους να πάνε πέραν της μάχης για να βρουν το δίκαιο τους πιο εύκολα από ότι αν παραμείνουν στο γαλλικό δίκαιο. Δεν έπρεπε να το πω εγώ, διότι ε, είμαι άντρας της συμβολεογράφος. Συνήθως ότι γλιτώνουν καλύτερα οι άντρες. Στην ε, Αγγλία, αν η σύζυγος που έχει βεβαίως την επιμέλεια των, η σύζυγος που επιμέλεια των παιδιών θα κρατήσει το σπίτι αν θέλετε, το οποίο μένει. Στη Γαλλία δεν είναι προφανή ε, αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν διαφορά στην νομοθεσία, γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά προηγουμένως. Σας ευχαριστώ για αυτές τις εξηγήσεις. Δεν θα συζητήσω σε αυτό που είπατε μεταξύ γυναικών και ανδρών, δεν είναι ο ρόλος μας. Θα δώσω όμως το λόγο στην κυρία Μπερζερό. Θα ήθελα να παρέμβω διότι ζω σε μια περιοχή στην οποία ζουν πάρα πολλοί Άγγλοι. Εγώ είμαι υπεύθυνη για κάποια θέματα τα οποία αφορούν τις δημοπρασίες και ε, μπορώ να πω ότι πολύ συχνά τα άτομα στα οποία αναφέρεστε είναι άτομα τα οποία μπορούν να επιλέξουν ένα γαλλικό δικαστήριο, Φερρυπίν και η γυναίκα να επιλέξει το αγγλικό δικαστήριο. Δεν είναι όμως πάντα έτσι τα πράγματα. Ε, πολλές φορές ε, χωρίζει κανείς ε, πηγαίνοντας στο δικαστήριο της περιοχής στην οποία είναι η ως τόπος διανομής του. Δεν ε, σκέφτεται πάντα να πάει να ζητήσει διαζύγιο στην Αγγλία. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ενώ έχουμε την, τα προγραμμιαία συμβόλαια, το 90% των Άγγλων τα αγνοούν. Αν λοιπόν γίνει εκ των προτέρων η επιλογή της διοικητικής αρχής μετά, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά, παρά το γεγονός ότι όπως ε, ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ισότητα σε αυτά τα θέματα μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και άλλων κοινοτικών χωρών. Πολύ καλά. Έχουμε χρόνο. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο και στον κύριο Τσέπελακ. Uh, Να συμπληρώσω λίγο την παρατήρησή σας για τα προβλήματα του δικαίου που υπάρχουν σε Ηνωμένο Βασίλειο και η περιοδική Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ε, κοινή περιουσία των συζύγων. Ήδη έχουμε πει ότι η λύση στο πρόβλημα θα ήταν να ενοποιηθεί η επιλογή των ε, κανόνων τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί ανεξάρτητα από το ποιο δικαστήριο θα αποτελέσει το αρμόδιο δικαστήριο τελικά. Θα εφαρμόσει το δικαστήριο αυτό όποιο και αν είναι τους ίδιους κανόνες για την επίλυση διαφορών οι οποίες θα οδηγήσουν στο ίδιο εφαρμοστέο δίκαιο. Και από όσο γνωρίζω εγώ, η τρέχουσα προπαρασκευαστική δουλειά που γίνεται για, την, για τον κανονισμό για το εφαρμοστέο δίκαιο, για τα καθεστώτα των ε, περιουσιών, ε, ακόμη. Οπότε αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια λύση. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα είναι αν τα βρετανικά δικαστήρια θέλουν να αναγνωρίσουν ε, τα ε, προγαμία συμβόλαια που συμφωνούν οι δύο σύζυγοι εάν το πράττουν. Και από όσο ξέρω, το, το κάνουν τα Βρετανικά δικαστήρια, τα αποδέχονται τέτοιου είδου συμβόλαια. Θέλουν, δείχνουν δηλαδή καλή θέληση ως προς αυτό, ότι η σύζυγος έχει συνάψει με μια, ένα προγραμμιό συμβόλαιο δυνάμει του γαλλικού δικαίου ας πούμε. Παρόλο που είναι περίπλοκο υπάρχουν κάποιες διέξοδοι ή εν υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, ας το πω έτσι καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Δεν ξέρω βέβαια ποια θα είναι αυτή η βελτίωση, αλλά Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κρόν και μπορείτε να φύγετε ελεύθερος όταν έρθει η ώρα. Να ακούσουμε τώρα την Κομισιόν. Ο κύριος Σότερ θα ξεκινήσει. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Ντελβό. Ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι εδώ για να μιλήσω για τον Βρυξέλλες 2α. Η τελευταία φορά που ήρθα ήταν το Φλεβάρι. Και αν δεν κάνω λάθος τότε είχαμε συζητήσει για τον κανονισμό 2α προς την ε, ε, αναθεώρηση. Τώρα η ακρόασή σας ε, έχει τίτλο «Η μεταρρύθμιση» του Βρυξέλλες 2α. Οπότε από, το, από τη δική σας την πλευρά τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Και θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς θα γίνουν και πιο συγκεκριμένα από την πλευρά τη δική μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που επικεντρωθήκατε σε αυτόν τον κανονισμό γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό μέσο για την ε, ζωή πολλών πολιτών. Έχουμε υπολογίσει ότι μιλούμε για περίπου 140.000 διεθνή ε, διαζύγια στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Είναι αρκετά υψηλό το νούμερο ε, κυρίως των ανθρώπων που επηρεάζονται από την περιπλοκότητα αυτή των ε, διασυνοριακών διαζυγίων και βεβαίως πέραν αυτού ε, επηρεάζονται και τα παιδιά που εμπλέκονται σε όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Αυτό λοιπόν το μέσο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημαντικό και για όλους εμάς να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Δράτω με τις ευκαιρίες, πριν σας ξεκινήσω για το που βρισκόμαστε και το πώς έχουμε προχωρήσει από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, τον ε, Φεβρουάριο, για να σας πω ότι η Κομισιόν δουλεύει πολύ σοβαρά προς την κατεύθυνση αυτή της μεταρρύθμισης του κανονισμού. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που μας ε, συμβουλεύουν για διάφορα θέματα νομικά και ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχει ακόμη μια συνάντηση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που θα γίνει. Επίσης, εσωτερικά, Έχουμε λάβει την πολιτική έγκριση να συνεχίσουμε προς την πρωτοβουλία αυτή της μεταρρύθμισης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό βήμα για εμάς στις εσωτερικές μας διαδικασίες δεδομένης και της σημασίας που αποδίδεται από την νέα Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διαδικασία της καλύτερης διακυβέρνησης. Ε, ως ξετμήμα αυτού, επειδή λοιπόν έχουμε αυτή την πολιτική έγκριση, καταφέραμε να δημοσιεύσουμε ένα, μια αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία έγινε, ε, δημοσιεύτηκε την προηγούμενη Παρασκευή, είναι online, είναι στο διαδίκτυο και είναι ένα κομμάτι της ε, ενισχυμένης δεσμεύσης της Κομισιόν να επιφέρει διαφάνεια στην νομοθετική διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν online αυτή η ε, αξιολόγηση δικτύπου και εκεί μπορείτε να δείτε τις διαφορετικές παραμέτρους, ε, τη όλες διαδικασία που γίνεται, τις διάφορες επιλογέ επιλογές πολιτικής που υπάρχουν. Υπάρχει η δυνατότητα των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού, όποιου θέλει δηλαδή, να κάνει σχόλια. Ε, δεν είναι ε, ε, δημόσια διαβούλευση αυτή καθ' αυτή, γιατί αυτή έγινε ήδη πέρσι, αλλά είναι ένα επιπλέον, μια επιπλέον δυνατότητα, πρωτοβουλία για να ανοίξει η διαδικασία αυτή στο κοινό, ώστε να τους δοθεί μια ακόμη ευκαιρία να πούν την άποψή τους. Και επίσης ε, μπορούμε ακόμα να συμπεριλάβουμε τα σχόλια των πολιτών στο, στη δουλειά μας. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει μια ε, ομάδα που με συναντήσεις ε, με εμπρογνωμόνε από τα κράτη-μέλη γιατί είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τη θέση των κρατών μελών για το θέμα αυτό, γιατί ούτως ή άλλως θα είναι φάκελος που θα πάει σε ομοφωνία, οπότε καλό θα ήταν να γνωρίζουμε οι μεν πολύ καλά τι πιστεύουν οι δε. Ε, και είναι, σήμερα μάλιστα είναι αυτή η συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες και γίνεται τώρα. Ε, επίσης, το Νοέμβριο θα γίνει μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου στο Λουξεμβούργο, η οποία θα αφιερωθεί στην αναθεώρηση αυτού του μέσου, που επίσης θα μας ε, δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία για να έχουμε στοιχεία από τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιούν τελικά αυτό το μέσο, από τους επαγγελματίες, τους νομικούς, τους συμβολεογράφους, Επίσης, οι δικαστικές αρχές και οι κεντρικές αρχές όλοι συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, οπότε θα είναι και αυτό μια πολύ καλή ε, ευκαιρία. Μετά από όλα αυτά, πρέπει να ξεκινήσουμε την εσωτερική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να γίνει αξιολόγηση αντικτύπου και έχουμε θέσει ως στόχο να γίνει αυτό εντός του τρέχοντος έτους. Αυτό θα μας διευκολύνει στις αρχές του 2016 να υποβάλλουμε την πρότασή μας, ελπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε η πρόταση αυτή να υποβληθεί το πρώτο εξάμεινο του 2016. Αυτά έτσι συνοπτικά για το πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά της υπόθεσης. Σε ό,τι αφορά τώρα το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε, Προφανώς δεν το επιλέξαμε τυχαία. Είδαμε ε, τα σχόλια που έχουν γίνει, τις ε, πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει εδώ το Φεβρουάριο, την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, μελέτη που παρουσιάστηκε εκεί. Επίσης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μία έκθεση τον Απρίλιο του 2014, η οποία επίσης δημοσιεύτηκε και έδειχνε έτσι, χοντρικά πού, πού υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθούμε, σε ποια σημεία αυτού του μέσου με βάση την αξιολόγηση που είχαμε κάνει. Ταυτόχρονα ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβούλευση το 2014, η οποία ε, ολοκληρώθηκε πέρσι το καλοκαίρι. Και όλα αυτά τα στοιχεία μας βοήθησαν να επικεντρωθούμε στους ε, τομείς κλειδιά για να προχωρήσουμε. Γενικώ είδαμε ότι ο κανονισμός αυτός είναι ένα πολύ καλό μέσο, ένα πολύ καλό εργαλείο, έχει προστιθέμενη αξία, πέραν του συστήματος της Σύμβασης Χάγης και λειτουργεί συνολικά καλά. Αλλά ε, υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να λειτουργεί καλύτερα. Και σε αυτούς ακριβώς πρέπει να επικεντρωθούμε. Η συζήτηση που μόλις κάναμε πριν πάρω το λόγο ήταν πραγματικά πολύ επίκαιρη σε ό,τι αφορά την ε, αυτονομία ό,τι αφορά την επιλογή που έχει κανείς, ε, την επιλογή δικαστηρίου και αυτή, η συζήτηση όντως, ε, ε, αυτό το θέμα έδωσε λαβή για αρκετά σημαντικά σχόλια. Σε έναν ιδιαίτερο κόσμο όλα τα κράτη-μέλη θα συμμετείχαν στην, στον κανονισμό Ρώμη 3, γιατί αυτό θα έδινε τη λύση ώστε να αποφύγουμε την, τον, την επίγουσα προσφυγή στα δικαστήρια. Η επιλογή του δικαστηρίου Μάλλον το κίνητρο για να, να φτάσει κανείς γρήγορα στο, στο δικαστήριο ε, ακυρώνει όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίως ξέρουμε ότι αυτό το θέμα είναι αρκετά δύσκολο. Είναι ένα θέμα που έπρεπε να ενταχθεί στο πρώτο, στο πρώτο, στο πρώτο τέτοιο νομικό κείμενο που είχαμε, το ΡΟΜΗ 3, και από κάποια κράτη-μέλη είχαμε σαφείς ε, απόψεις προς αυτό, αλλά όχι από όλα φαντάζομαι ότι και στο προβλεπόμενο μέλλον ε, έτσι θα γίνει. Δεν πρόκειται να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό σε τούτη τη μεταρρύθμιση, ούτε έχουμε ως στόχο να το κάνουμε. Βεβαίως, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε όποιον θέλει να ενταχθεί στον ε, κανονισμό ορομετρία. Αυτό όμως που θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο ως έτσι, στοχευμένη βελτίωση θα ήταν η δυνατότητα να παράσχουμε στους συζύγους τη δυνατότητα και βέβαια ε, ο μιλητής πιο πριν είπε ότι δεν θα γίνεται σε κάθε περίπτωση και είναι σωστό, αλλά σε κάθε περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμο αν λοιπόν οι σύζυγοι είχαν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν, να καταλήξουν σε μια τέτοια συμφωνία ανάλογα με την εθνικότητα ας πούμε, πάλι στα πλαίσια της ε, αυτονομίας των μερών, έτσι ώστε να υπάρχει σαφήνεια, διαφάνεια, για να ε, ευθυγραμμίσουμε λιγάκι και το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσει στα πλαίσια του Βρυξέλλες 2α. Ε, σε σχέση και με εργαλεία που έχουμε από, με ε, νομικά κείμενα που έχουμε όπως ας πούμε ο κανονισμός για τις διατροφές. Οπότε θα πρέπει μάλλον να υπάρξει ένας μικρός βαθμός έστω αυτονομίας των μερών ώστε να μπορούν οι σύζυγοι να επιλέγουν το δικαστήριο. Και αυτό βεβαίως θα δώσει και κάποια πλεονεκτήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τις διάφορες διαδικασίες, στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό και δυνατό βεβαίως, σε μία. Και όλε αυτέ θα τι αναλαμβάνει μία δικαιοδοσία, μία δικαστική αρχή. Τώρα, για τα θέματα που αφορούν στα παιδιά, που είναι βεβαίω πολύ ευαίσθητο τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ προσεκτική στο να εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα και βεβαίως προ το συμφέρον του παιδιού. Άλλος ένας στόχος που έχουμε θέσει και είναι πολύ σημαντικός είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όλα αυτά τα θέματα η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, το συμφέρον του παιδιού, ε, η αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη συνδέονται. Είναι ο μπούσουλα που ε, ξεκινά και ολοκληρώνει την όλη διαδικασία μεταρρύθμιση. Θα μπορούσα να σα δώσω βέβαια και κάποια παραδείγματα αναφερόμενο σε συγκεκριμένε ιδέε που έχουμε σκεφτόμαστε κάποια περαιτέρω βήματα για να ακυρώσουμε πια την, αυτή την τυπικότητα του εξεκουάτουρ. Ο κανονισμός 2α, Βρυξέλλες 2α, ήδη έχει κάνει κάποια βήματα ως προς αυτό, αλλά στα ό,τι αφορά την ε, επιμέλεια ε, δεν ήρθε στο ύψος των ε, περιστάσεων. Οπότε γι' αυτό θέλουμε να ακυρώσουμε, να υπάρξει ανάκληση του εξεκουάτου. Σε ό,τι αφορά τώρα την αδιατύπωση του Βρυξέλλες 2α, θέλουμε να, να εξαλειφθούν τέτοιες τυπικότητες που δεν βοηθούν, που ίσως να είναι και επιβαρυντικές για τα μέρη. Ακριβώς στα πλαίσια του κανονισμού 2α και κυρίως γι' αυτόν επειδή εμπλέκονται και παιδιά. Όπου εμπλέκονται παιδιά έχουμε έναν λόγο παραπάνω να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε αποτελεσματικοί και ταχείς. Γιατί ο χρόνος έχει σημασία. Και έχει πραγματικά ε, πολύ σημαντικές ε, συνέπειες στα παιδιά. Ό,τι λοιπόν υπάρχει, όταν υπάρχουν ε, προβλήματα που εμποδίζουν την γρήγορη διεξαγωγή τέτοιων υποθέσεων θα πρέπει να τα δούμε. Επίσης, βλέπω ο κύριος Βεύκα είναι εδώ και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με το Βρυξέλλες 2α Μπορούμε λοιπόν να εμπνευστούμε από όλα αυτά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παλιά μας εμπειρία. Δεν δεν, το θέμα δεν είναι μόνο οι δικλείδες ασφαλείας, ε, χρειαζόμαστε και μάλλον θα χρειαστούμε και πολύ περισσότερες, κυρίως όταν μιλάμε για τα παιδιά. Αλλά η συστηματική αυτή τυπικότητα που είναι το εξακουάτος, που εφαρμόζεται σε μια φάση εξάντε, θα μπορούσαμε να το καταργήσουμε για να υπάρχει ελεύθερη ροή αποφάσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές, στα πλαίσια βεβαίως της ε, αναδιατύπωσης, οι οποίες μπορούν να ακυρωθούν από τα μέρη εάν θεωρήσουν ότι έχει υπάρξει κάποια παρατυπία στην όλη διαδικασία ή αν δεν ε, είχαν, αν δεν έλαβαν τα συνοδευτικά έγγραφα, τα εισαγωγικά έγγραφα της δίκης ή οτιδήποτε. Ή αν δεν, το παιδί δεν έχει πει την άποψή του, δεν έχει παραστεί σε ακρόαση. Ένας από τους λόγους λοιπόν, ένας ακόμα από τους λόγους που θέλουμε να καταργήσουμε το εξεκουάτρο. Επίση, Επίσης, η ευθυγράμμιση των διαδικασιών. Για την εκτέλεση, ακόμα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες κολλούν, μπλοκάρονται είναι μια πολυτέλεια την οποία δεν έχουμε και πρέπει να σταματήσει αυτό. Εδώ έρχεται να παίξει ρόλο η αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη. Υπάρχουν υποθέσεις που μπλοκάρονται όταν δεν υπάρχει επιτόπου εκτέλεση. Και βεβαίως διαβρώνεται και η αμοιβαία εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να υπάρξει αυτή η ταχεία διεξαγωγή και εκτέλεση του μέσου. Οπότε παρόλο που είναι δύσκολος αυτός ο τομέας της εκτέλεσης, το αναγνωρίζω σαφώς, Πρέπει να είμαστε πολύ επικοδομητικοί και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή θα βελτιωθεί επιτόπου. Σαφώς και δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το δούμε για να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Επίσης, άλλο ένα δύσκολο ζήτημα ήταν η ακρόαση, είναι η ακρόαση των, των παιδιών στο δικαστήριο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ρυθμίζουν διαφορετικά τα κράτη-μέλη. Όλα τα κρατημέλη όμως έχουν ε, ε, συνυπογράψει την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Γιατί, πιστεύει ότι όλα, ε, γιατί δείχνει ότι όλα τα κρατημέλη έχουν αποδεχτεί αυτές τις υποχρεώσεις. Τούτου λεχθέντος, Βεβαίω έχουν υπογράψει ακριβώ λόγω και τη αυτονομία που του δίνει αυτό, αλλά έχουν τελείω διαφορετικέ διαδικασίε για το πώ γίνεται, πώ ε, διεξάγεται η ακρόαση ενό παιδιού. Αυτό που πρέπει εμεί να διασφαλίσουμε είναι ότι αυτέ οι διαφορέ δεν θα εμποδίσουν την ελεύθερη ροή διακίνηση των αποφάσεων. Και αυτό πρέπει να γίνει με έναν ευαίσθητο, εύλογο τρόπο. Πρέπει να δούμε τι είναι απαραίτητο πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε λίγο αυτές τις ε, αποφάσεις των ε, δικαστηρίων και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη σε αυτό το τομέα, στο πώς δηλαδή θα διεξάγεται η ακρόαση των παιδιών. Δεν είναι εύκολο και το μελετούμε πολύ προσεκτικά για να δούμε ποιος είναι ο πιο καλός τρόπος, ποιος, ποιο είναι το καταλληλότερο επίπεδο παρέμβασης που θα πρέπει να έχουμε. Γιατί βεβαίως είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι, αυτές είναι κάποιες πτυχές ε, ε, του σκεπτικού μας. Επίσης, άλλος ένα σημαντικός τομέας, ε, τον οποίο τον συζητήσαμε και το Φεβρουάριο, είναι το θέμα της απαγωγής παιδιών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του μέσου αυτού και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο υπάρχον στόχος του άρθρου 11 θα λειτουργήσει όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται. Το άρθρο 11 έχει στόχο να εξασφαλίσει την ε, ταχεία επιστροφή ενός απαχθέντος παιδιού στη χώρα προέλευσής του. Ε, αυτό θεωρούμε ότι γενικώ λειτουργεί καλά, αλλά και πάλι υπάρχουν κάποιες επιμέρους περιπτώσεις που ε, μας δείχνουν ότι δεν λειτουργεί τελικά όσο καλά θα έπρεπε. Μελετήσαμε λοιπόν το τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της διαδικασίας του άρθρου 11 στα πλαίσια αυτού του κανονισμού και νομίζω ότι αντί να προτιμήσουμε μια ε, ε, ραγδαία αλλαγή του 11 να κάνουμε μια πιο στοχευμένη ε, τροποποίησή του. Ας πούμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το, αυτή την προθεσμία των 6 εβδομάδων που υπάρχει. Οι 6 εβδομάδες υπάρχουν, έχουν κάποια πλέον εκτήματα, θέτει βεβαίως έναν πολύ φιλόδοξο στόχο, δίνει ένα σαφές μήνυμα ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο φιλόδοξη που σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται. Οπότε πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε καλύτερα ότι θα επιστρέψει άμεσα το παιδί. Άλλη μία δυνατότητα είναι να δούμε, επειδή σε πολλά ε, κράτη-μέλη βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες διαδικασίες έφεσης, μετά μια δεύτερη, μια προσφυγή ακόμη, θα πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό προσφυγών που επιτρέπονται στα πλαίσια αυτά δεδομένου το ότι ο κανονισμός δίνει αυτή την ε, προθεσμία των 6 εβδομάδων. Ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, αυτό δεν τηρείται καθόλου. Οπότε μήπως θα πρέπει να διορθώσουμε ίσως τον αριθμό των δυνατοτήτων προσφυγής. Άλλο ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι αν πρέπει να αλλάξουμε τις, τον, την ανασταλτική ε, λειτουργία αυτού του κανόνα. Υπάρχουν εξειδικευμένα δικαστήρια σε πολλά κράτη-μέλη που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτή την εξειδικευμένη διαδικασία. Ξέρουν τους ε, ομολόγους τους και σε άλλες ε, χώρες, σε άλλα δικαστικά συστήματα και αυτή η φιλική ας πούμε σχέση, η οικειότητα βελτιώνει τη λειτουργία του εργαλείου. Οπότε καλό θα ήταν να δούμε και το θέμα της συγκέντρωσης της, αρμο... της δικαιοδοσίας. Επίσης υπάρχει μια δυνατότητα το δικαστήριο να εξασφαλίσει ότι θα επιστραφεί το παιδί στο δικαστήριο της χώρας κατα, καταγωγής όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πάντα, δεν είναι σαφές, δεν, ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει ε, να τηρούνται όλοι οι κανόνες και να υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις. Άλλος ένας ε, παράγοντος που είναι επίσης σημαντικός είναι η διευκόλυνση της δουλειάς των αρμοδίων αρχών, των κεντρικών αρχών. Έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στην καθημερινή εφαρμογή του κανονισμού. Αλλά και στα πλαίσια της διαδικασίας επαγωγής παιδιού. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των κεντρικών αρχών. Επίσης, άλλος ένας πιθανός περιορισμός που μελετούμε και θέλουμε να βελτιώσουμε είναι το ότι προς το παρόν τα, μέτρα που λαμβάνονται, τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται από το τελικό δικαστήριο περιορίζονται στη δική του δικαιοδοσία και δεν έχουν, ε, ε, ε, δεν έχουν επίδραση πέραν της δικαιοδοσίας αυτού. Κατανοώ βεβαίω τη θέληση του δικαστηρίου του τελικού να επιστρέψει το παιδί στο δικαστήριο καταγωγής, της χώρας καταγωγής, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο, στο δικαστήριο καταγωγή, υπάρχουν κάποιε διαδικασίε οι οποίε προστατεύουν, α πούμε, το παιδί για μία-δύο εβδομάδε μέχρι το δικαστήριο καταγωγή να ξαναδικάσει ε, την υπόθεση. Και αυτό θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμο στη χώρα καταγωγή. Αυτό προ το παρόν δεν γίνεται. Θα μπορούσε όμω να διευκολύνει την. Ε, το δικαστήριο το τελικό να επιστρέψει το παιδί στη χώρα καταγωγής εάν εξασφαλιστεί ότι θα μπορούσε μέσα σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα το παιδί να προστατεύεται με κάποιες συγκεκριμένε δικλείδες. Μπορώ να συνεχίζω για πολλή ώρα. Ε, υπάρχουν ε, πολλά, πολλά σημεία που είναι αρκετά πρακτικά και νομικά βεβαίως για τα, και τα οποία θέλουμε να αλλάξουμε για να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε την διαδικασία του άρθρου 11 του κανονισμού. Και το τελευταίο ζήτημα που ήθελα να τονίσω, γιατί είναι και αυτός ένα σημαντικός τομέας, είναι η συνεργασία γενικών των κεντρικών αρχών. Όχι μόνο στα πλαίσια του άρθρου 11, γιατί αυτό είναι το μηχανοστάσιο ουσιαστικά του κανονισμού. Είναι το πώς οι αρχές λειτουργούν η μία με την άλλη, πώς συνεργάζονται. Βλέπουμε ότι στο άρθρο 55 του Βρυξέλλες 2α να περιλαμβάνει κάποια στοιχεία, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο σαφές για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό που ορίζει στην πράξη. Καλύτερη δηλαδή ε, σαφήνεια, καλύτερη διαφάνεια στη διατύπωση του 55, που θα μπορούσε να βελτιώσει πραγματικά την καθημερινή δουλειά των κεντρικών αρχών. Οπότε το μελετούμε και αυτό. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνάντηση ε, στις αρχές του Νοέμβρη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, γιατί εκεί θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί εκεί θα μιλήσουμε με τις κεντρικές αρχές. Επίσης, ένα τμήμα αυτού έχει να κάνει και με τη συνεργασία ε, στα πλαίσια του άρθρου 56 του κανονισμού, που αφορά στην ε, τοποθέτηση του παιδιού σε ε, θετές οικογένειες. Αυτή η διάταξη δεν λειτουργεί πάντα όσο καλά θα έπρεπε. Είναι βεβαίω αρκετά ευαίσθητο το θέμα γιατί μια κεντρική αρχή καμιά φορά δεν καταλαβαίνει επακριβώ τι κάνει μια άλλη αρμόδια κεντρική αρχή ε, και τα, πολλές φορές οι θετές οικογένειες και τα παιδιά βρίσκονται σε διαφορετική ε, σε διαφορετική δικαιοδοσία και ε, είναι δύσκολο να οριστεί η αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Διέτρεξα σχετικά γρήγορα όλες αυτές τις ε, πτυχές. Η Τζοάννα δίπλα μου τα ξέρει πολύ καλύτερα, πολύ λεπτομερέστερα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστω να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Σάτας. Η κυρία Ζαντίσκαν δεν θα μιλήσει τώρα, θα μιλήσει. Όχι, όχι, δεν θα μιλήσει. Η κυρία Μακίνας έχει καθυστερήσει. Φαντάζομαι ότι θα έρθει σε κανένα τέταρτο. Εγώ θα ε, έλεγα να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Τσιάφκα, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις τόσο ενδιαφέρουσες προκατακτικές παρατηρήσεις που έχουν σχέση με την αναθεώρηση του Βρυξέλλες 1 και 2. Θα συζητήσουμε εκτενώς για τα, τις διάφορες πτυχές αυτής της αναθεώρησης. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν εργάστηκα για το Βρυξέλλες 1, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξάρτηση του κανόνα εξετουάτων, αρχικά φαινόταν ένα άθλος. Και είχα το φόβο ότι η διαδικασία αυτή θα έπρεπε να διαρκέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι ο κανονισμός αυτός αφορά ιδιαίτερα τον επιχειρηματικό κόσμο. Τώρα εδώ μιλάμε για προβλήματα που αφορούν ένα συγκεκριμένο άτομο. Ένα άτομο που βλέπει να διαλύεται ο γάμος του και βλέπει και ένα παιδί που υποφέρει. Θα πρέπει συνεπώς να κάνουμε μερικές αλλαγές, αλλά με προσοχή. γιατί αυτό επηρεάζει ανθρώπινες ζωές. Και οι Βρυξέλλες 2 ε, και η Ρώμη 1 μας δείχνουν ότι κρύβονται πάρα πολλές δυσκολίες πίσω από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Για παράδειγμα, εμείς λέμε ε, πώς θα πρέπει να ακούγεται μια διάταξη. Η δική μου εμπειρία από τότε που ετέθη σε το Βρυξέλλες 1 μετά τις τροποποιήσεις του μου δείχνει ότι η άγνοια αυτό που θα πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες συνεχίζει να παραμένει πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή πάρα πολλές φορές είναι άγνωστα αυτά που καλούμε, θα, ή καλούνται να εφαρμόσουν με δυσαρέστησε πάρα πολύ ο κανονισμός ε, Ρώμη 3 επί του οποίου εργάστηκα ως εισηγητής. δώσαμε στα ζευγάρια ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα την επιλογή του αρμόδιου δικαστηρίου σε περίπτωση διαζυγίου. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και στις Εξέλες 2. Σκέφτομαι και το θέμα της προστασίας του παιδιού σε κάθε περίπτωση ο κανονισμός αυτός για τον οποίο μιλάω δεν έγινε δεκτός από όλα τα κράτη-μέλη. Για πρώτη φορά στην ιστορία επιλέξαμε μία διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας και ενδεχομένως αυτό είναι το μοναδικό πλεονέκτημα. Αυτή η λύση όμως θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες μέλη γιατί αυτό θα διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στην προηγούμενη ιδέα. Η συνθήκη εκ των νου είναι η αρμόδι να είναι ε, γνώστες αυτών των, δυνατοτήτων. Το σημαντικό είναι ότι οι τελικοί χρήστες να γνωρίζουν και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Το ίδιο να συμβαίνει και με τους υπεύθυνου που θα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Έχω λοιπόν ένα φόβο γιατί επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στους διάφορους κανόνες που θα πρέπει να τροποποιηθούν για να μπορέσουμε να τους απλοποιήσουμε. Το δεύτερο αυτό μέρος που αφορά την υποχρέωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών μελών να ελέγξουν την εφαρμογή του κανονισμού είναι κάτι που τίνουμε να ξεχνάμε. εσείς σας παρακαλώ, πόσα άτομα πηγαίνουν στο Λουξεμβούργο. Είναι άτομα ενημερωμένα, είναι άτομα που ενδιαφέρονται. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να έπαιρναν μέρος περισσότεροι άνθρωποι σε αυτές τις συνεδριάσεις. Θα μπορούσαμε να στραφούμε στα εξειδικευμένα τμήματα των δικαστηρίων, δηλαδή αυτά που ασχολούνται με το οικογενειακό δίκαιο. Τώρα σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των δικαστών και πάλι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα που επιβραδύνουν την εισαγωγή αυτών των διατάξεων. Εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η συνεργασία που μας περιμένει. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όλοι και οι δικαστές και οι αρχές που είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή του νόμου και οι τελικοί χρήστες θα βρίσκονται στο κέντρο των εργασιών μας. Και θα ήθελα μεταξύ των άλλων να υπογραμμίσω το θέμα του καλού του παιδιού. Τι είναι προς όφελος του παιδιού. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Ε, γιατί ε, ε, είναι μια ιστορία το τι κάνουν οι ενήλικες με τη ζωή τους. Τα παιδιά όμως θα πρέπει να έχουν κάθε προστασία σε ό,τι αφορά ε, τα περιουσιακά του στοιχεία και, τις, ε, και τα, δικαιώματά τους. Πιστεύω ότι αυτό, αυτή είναι η πηξίδα που θα πρέπει να μας ε, καθοδηγεί βεβαίως. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσέγγισης στις διάφορες χώρες. Δεν θέλω να μιλήσω για τις ε, ανάδοχες οικογένειες που νομίζω θα πρέπει να βγουν κατά μέρος. Είναι θέματα όπως η οθεσία που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις που τα εθνικά δικαστήρια παραπέμπουν τα θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Και δίχως άλλο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα διότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες παρέμβασης και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η βάση την οποία διαθέτουμε για να βελτιωθούμε, αλλά όπως ξέρουμε θα πρέπει να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για να βελτιωθεί η κατάσταση κυρίως για θέματα ευημερία των παιδιών, το οποίο δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για όλες τις παρουσιάσεις και τις εξηγήσει που δώσατε, γιατί βλέπουμε ποια είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί για την θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Τσέφκα. Σωστά είπατε όντως ότι το πρωταρχικό θέμα που μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό συμφέρον του παιδιού. Αυτό είναι ο πρώτος αντικειμενικός στόχος της καθημερινότητάς μας. Επίσης, ε, ε, συμφωνώ και σημειώνω αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να κάνουμε ευφυείς, έξυπνες αλλαγές και θα πρέπει να μπορέσουμε να περάσουμε από τους τομείς τους οποίους είναι καλοί κανόνες αλλά ίσως δεν λειτουργούν τόσο καλά όσο θα έπρεπε γιατί δεν υπάρχει απόλυτη ε, συνειδητοποίηση. Θα πρέπει περισσότερη ενημέρωση να έχουν και οι πολίτες και αυτοί που πρέπει να τους εφαρμόσουν και να περάσουμε κυρίως σε αλλαγές για θέματα λειτουργίας, σωστής λειτουργίας του όλου μέσου αυτό που διαθέτουμε. Το συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν έχουμε νέους βελτιωμένους κανόνες, θα πρέπει να τους κοινοποιήσουμε στα, στον κόσμο, να τους ανακοινώσουμε. Συνειδητοποιούμε το γεγονό ε, ότι ο καλύτερος κανονισμός ε, του, του κόσμου θα μπορούσε να είναι η νέας κανονισμός των Βρυξελών, αλλά εάν δεν ενημερώσουμε τον κόσμο, δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέγω ότι είναι το δίκτυο αυτό το οποίο προανέφερα πάρα πολύ σημαντικό διότι μπορεί να ενεργήσει ως πολλαπλασιαστής και να μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα νομοθετικά όρια στα οποία συζητούμε όταν κάνουμε αλλαγές στην νομοθεσία, στις νομοθετικές πράξεις και να περάσουμε στην πράξη. Έχουμε λοιπόν μια συνάντηση για τον κανονισμό 1 Βρυξελών αυτή την ε, Παρασκευή για να συζητήσουμε συγκεκριμένα το θέμα αυτό της, uh, uh, της αναδιατύπωσης του, ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Σωστά λοιπόν αναφέρατε αυτά τα που είπατε. Ακόμη και με τα θέματα τα οποία αφορούν τα θέματα ε, κληρονομιάς. Και συνειδητοποιήσαμε ότι εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μέσο στο διαθεσί μας, αλλά και το καλύτερο του κόσμου να ήταν, αν δεν το γνωρίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να επιτύχει. Κάναμε λοιπόν μία εκστρατεία κοινοποίησης του, διαφήμισής του αν θέλετε, ε, αυτού του συνόλου κανόνων που αφορά τη κληρονομιά στο καλοκαίρι και είδαμε ότι πραγματικά από το feedback που είχαμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πρέπει το γνωρίζει ο κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα με τι παρατηρήσει που κάνατε και για την ανάγκη ότι όντω θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα σε θέματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν και να γίνουν πιο ορθολογικά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά κανένας άλλος συνάδελφος το λόγο. Και θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Σωστά κατάλαβα ότι αστιάζεστε περισσότερο στα θέματα που αφορούν τα παιδιά παρά σε άλλα θέματα που αφορούν τα διαζύγια. Για θέματα που αφορούν τον γάμο και τις διαφορές που μπορούν να προκύψουν, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, αν θέλετε για τέτοια θέματα η συνάδελφος μπορεί να σας ενημερώσει. Αλλά γενικά Πρέπει να πω ότι το κύριο μέρος των εργασιών μας αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με τα παιδιά. Η συνεργασία την οποία προανέφερα τα διάφορα άρθρα αφορούν αποκλειστικά τα θέματα που αφορούν τα παιδιά. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να αλλάξουμε για τα άλλα θέματα των διαφορών στο γάμο. Η μπορεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Ε, και εμεί ε, συζητάμε θέματα που κατά την άποψή μα είναι σημαντικά για τα ζευγάρια όταν λάβουμε υπόψη μας την όλη κινητικότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μία μελέτη του Κοινοβουλίου αναφέρει ότι υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις διαζυγίου και χωρισμού. Ενδεχομένω πρέπει να υπάρχει ένα δικαστήριο που να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες αυτοί να υποβάλουν το αίτημά τους. Για την ώρα είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Εάν η συνήθις κατοικία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι δύσκολο να υποβάλλεται το, το αίτημα. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχει κάποια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρξει τέτοια δυνατότητα. Τώρα, η άλλη περίπτωση αυτό αφορά όταν υπάρχουν εκρεμή οικογενειακά ζητήματα, ας πούμε θέματα γονικής μέρημνας. Θα μπορούσατε να έχετε άλλες εκκρεμότητες ή τις ίδιες εκτεμότητες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε αυτό το ζευγάρι. Στο τέλος θα πρέπει να ληφθούν δύο αποφάσεις και οι αποφάσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι διαφορετικέ. Όπως αναφέρθηκε σε ένα κανονισμό θα μπορούσε να υπάρχει κάποια ελαστικότητα στον δικαστή καταρχάς για να αναστείλει ε, τη δίκη να δει εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφασίσει εάν θα, γίνει, θα αναγνωστεί αυτή η απόφαση από το εξωτερικό ή να συνεχιστεί η δίκη η οποία είχε ε, διακοπεί. Αυτά είναι θέματα που λαμβάνουμε τώρα υπόψη μας και αυτό σε θέματα που ε, αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις. Ευχαριστώ. Ah. Uh, uh, η κυρία Μαγκίνες μόλις προσγειώθηκε. Δεν ξέρω πού ακριβώς όμως. Καθυστέρησε η πτήση της, οπότε μάλλον δεν θα έρθει σήμερα. Δεν ξέρω, ίσως να μπορέσει να μας στείλει την παρουσίασή της, να μας ε, την καλέσουμε κάποια άλλη φορά. Εν πάση σήμερα δεν θα την ακούσουμε πάντως. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπελακ. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα, παρακαλώ να πω κάτι. Μιλούμε για ε, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την γονική μέρημνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός επιστροφής ενός παιδιού που υπάρχει στον Βρυξέλλες 2α ουσιαστικά είναι μία προσθήκη στην ε, συνθήκη της Χάγης και η σύμβαση της Χάγης εφαρμόζεται και μεταξύ οποιασδήποτε άλλης χώρας, όχι μόνο ευρωπαϊκής, που τη δεσμεύει αυτή η σύμβαση. Οπότε σε ένα βαθμό ο κανονισμός αυτός ε, ε υπερέχει της, ε, του Βρυξέλλες 2, ο 1374 2000 πρώην ε, Βρυξέλλες 2 του 2000. Ε, αυτός ο μηχανισμός λοιπόν εφαρμόζεται εντός των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσο πιο πολύ εφαρμόζεται εντός της Ένωσης τόσο πιο ασυμβίβαστος είναι με το μηχανισμό που υπάρχει στον, στη Σύμβαση της Χάγης μεταξύ Αυστρίας, Ρωσίας ή Γερμανίας, Ελβετίας για παράδειγμα. Οπότε ρωτώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σχέδιο έχει στα πλαίσια, απέναντι στην, στην Σύμβαση της Χάγης. Σε ποιο βαθμό σκέφτεστε να αναθεωρήσετε αυτό το μηχανισμό που ε, υπάρχει στην Σύμβαση για να μην υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ των δύο γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο το θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν και οι υποχρεώσεις από τη συνθήκη ενός κράτου μέλους έναντι μιας τρίτης χώρας, οι οποίες διασφαλίζονται ακριβώς από την ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε σε ποιο βαθμό μπορείτε να εξυγχρονίσετε αλλά να είσαστε σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις που έχετε από τη συνθήκη. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Παρακαλώ. Σας ακούμε κύριε Σότερ. Καλωσορίζω πάντα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Το αν θα μπορέσω να σα απαντήσω επαρκώ είναι άλλο θέμα. Βεβαίω θα κάνω ό,τι μπορώ. Έχετε δίκιο. Ο Βρυξέλλες 2 ε, βασίζεται ουσιαστικά στην εμπειρία που υπάρχει και στην καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα στα πλαίσια της Σύμβασης της Χάγης. Τούτου λεφθέντος, όταν ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α υιοθετήθηκε, είδα, ήδη Είχαμε, ήδη έχω ένα ερώτημα, ένα, μια απάντηση για το ερώτημά σας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα της Χάκης είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό σύστημα συνεργασίας. Μεταξύ των κρατών μελών, ωστόσο, υπήρχε ήδη μια πολιτική βούληση να κάνουμε κάτι καλύτερο. Όχι για να υπονομεύσουμε την καλή λειτουργία του συστήματος, αλλά για να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι στο άρθρο 11 ας πούμε προστίθενται διάφορα στοιχεία για να ξεκαθαριστούν, για να βελτιωθούν τα όσα προβλέπονται, για να πάμε πιο μακριά, πιο μακριά από όσα θα μας επέτρεπε να πάμε ως η Σύμβαση της Χάγης. Και ουσιαστικά δεν θέλουμε να φύγουμε εντελώς, να απομακρυνθούμε από αυτή την ε, φιλοσοφία, γιατί το σύστημα της Χάγης είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ καλό και έχετε δίκιο, τα δύο συστήματα θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα οι δικαστές που γνωρίζουν τη σύμβαση της Χάγης δεν χρειάζεται να, δεν θα πρέπει να δυσκολεύονται πολύ να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες. Αν τώρα το, το σύστημα είναι δύσκολο, είναι πιο περίπλοκο, ναι, προφανώ είναι δύσκολο να εφαρμόσουν οι δικαστέ ε, τα δύο αυτά συστήματα, του δύο μηχανισμού. Τούτου λεχθέντο, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Έχουμε την κοινοτική μα μέθοδο που μα επιτρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα και να βελτιώσουμε τα σημεία όπου θέλ, χρειάζονται βελτίωση. Ενώ καμιά φορά στα πλαίσια τη Χάγη αυτό είναι λίγο δύσκολο. Οπότε γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία που μα δίνει, αυτή την ευκαιρία που μα δίνει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί αυτού πρόκειται. Δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε εντελώ από το σύμβαση τη Χάγη, ούτε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που δεν θα λειτουργεί καθόλου ε, με τη σύμβαση, με το μηχανισμό τη σύμβαση. Δεν θέλω καθόλου να έχετε αυτή την εντύπωση. Ευχαριστώ. Σα ικανοποίησε η απάντηση. Ε, ε, με ενθουσίασε μόνο, με ικανοποίησε η απάντηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίαση, για τη συζήτηση. Καλή τύχη σας εύχομαι, Κομισιόν. Μακάρι να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά μπορεί αυτός ο φάκελος. Και κάνουμε ένα διάλειμμα ως τις 5. Α, οκ, ε, και κλεισμένα των θυρών λοιπόν η συνέχεια. Σας ευχαριστώ όλους και θα τα ξαναπούμε στις 5.